Λοιπόν, σας προτείνω αγαπητοί συνάδελφοι να ξαναρχίσουμε. Στο 1.16 θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Όλε Κρίστενσεν για να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του, γνωμοδότησης καλύτερα, με θέμα τροποποίηση της οδηγίας 2008 106 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση στο ναυτικό. Εμείς νομοδοτούμε. Καθήλυνα αρμόδια είναι προφανώς η Επιτροπή Μεταφορών. Και εισηγητής, ο πρόεδρος αυτής, ο κύριος Μπράιαν Σίμψον. Ζητήσαμε εμείς να συνδεθούμε με αυτό το θέμα. Ε, και είχαμε διάφορες επαφές και συναντήσεις και δεν νομίζω ότι είναι θέμα άρθρου 50 σε αυτό. με την επιφύλαξη της τελικής ε, απόφασης για αυτό το θέμα, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό προτείνω να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε ότι είναι μια έκθεση αυτή άκρος τεχνική. Θα προσπαθήσω ε, να σας εξηγήσω σύντομα είναι μια σύμβαση STCW που έχει να κάνει με τους ναυτικούς και τα πληρώματα. Υπάρχει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός που εμπλέκεται εκεί, ο IMO, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά, εμείς ε, ανταποκρινόμαστε στις διεθνείς συμβάσεις και το 1978 εκρίθηκε και ε, το 2008 τροποποιήθηκε. Το 2007 ε, έγινε μια ε, επανεξέταση, ένας έλεγχος αυτών ε, των διατάξεων ε, για να δουν αν χρειάζεται τροποποίηση και ομόφωνα πλέον στη Μανίλα στις 25 Ιουνίου του 2010 αποφασίστηκε να ε, γίνει αυτή η τροποποίηση. Όλα αυτά που αποφασίστηκαν τότε τέθηκαν σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2011, 12, συγγνώμη. Εμείς λοιπόν τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και αν δεν μεταφερθεί αυτό και δεν μεταφερθεί στο κοινοτικό και στο εθνικό δίκαιο θα παραβιάζουν τα κράτη-μέλη διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, πρέπει να δράσουμε. Τα κράτη-μέλη είχαν την ευκαιρία τον Ιούλιο του 2011 να δουν την απόφαση και να αντιδράσουν, αλλά κανένα κράτος μέλος δεν αντέδρασε. Η παρούσα γνωμοδότηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι νέες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταποκρίνονται στην ισχύουσα κείμενη διεθνή τάξη και νομοθεσία και ε, θα ανταποκρίνονται σε υφιστάμενες συμφωνίες ε, για τα κοινωνικά. Στην έκθεση αυτή λοιπόν δεν γράφει τίποτα που να το έχω εφεύρει εγώ. Δεν, όλα είναι κείμενο δίκαιο. Εγώ δεν κάνω παρά μία διευκρίνηση στη γνωμοδότησή μου. Έχουμε μια σειρά λοιπόν διευκρινήσεων και επεξηγήσεων που από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφερόταν κάθε φορά η εκάστοτε οδηγία και κληθήκαμε εμεί να το κάνουμε, τονίσαμε και το ε, ρόλο των κοινωνικών εταίρων και σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης. Ξέρετε ότι είναι μια οδηγία του 99, υπαριθμόν 63 τότε, περί χρόνων εργασίας των ναυτικών. Και υπάρχουν και κάποια πιστοποιητικά. Είναι τεχνική οδηγία. Και φυσικά εδώ ισχύει και η ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Και εκτός από αυτές τις τροποποίησεις έχουμε και μια σειρά γλωσσικών αλλαγών. 6-7 τροπολογίες μας έχουν αυτό το στόχο, γλωσσική διόρθωση. Δεν ξέρω αν θα τις δηλώσουμε, αν θα τις ψηφίσουμε. Τώρα τα γλωσσικά έχουν να κάνουν με το φύλλο, άνδρας, γυναίκα. Στην Δανία έχουμε μια ουδέτερη έκφραση για το φύλλο και δεν χρειάζεται να διευκρινίζουμε κάθε φορά. Αυτά. Είναι λοιπόν τεχνική η γνωμοδότηση. Και σας είπα, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε και να προσαρμοστούμε και να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, Βεβαίω είμαι και σε επαφή με την καθήλυν αρμόδια Επιτροπή Μεταφορών. Δεν έχουμε εδώ διευρυμένη συνεργασία, δεν είναι το άρθρο 50, το είπε και η Πρόεδρος προηγουμένως. Εμείς θα αποφασίσουμε αυτά που μας αφορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή Μεταφορών να τα υιοθετήσει. Από τις επαφές που είχαμε την Επιτροπή Μεταφορών δεν ε, διαφωνούν με τίποτα. Χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, δεν είναι αντίθετη με αυτά που λέγω εγώ, είμαστε σε σενή επαφή. Και ελπίζω να μας λάβουν υπόψη. Το συζητήσαμε και με τους σκιώδεις ηγητές και ελπίζω το κείμενο αυτό να ευδοκιμήσει και να υποστηριχθεί για να μπορέσουμε να το στείλουμε στην Επιτροπή ε, Μεταφορών και να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διεθνείς συμφωνίες. Περιμένω με μεγάλη χαρά τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Ε, να e, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιγητή, τον κύριο Κρίστενσεν, για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε και για την προσήλωσή του στο θέμα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω πως όλες αυτές οι εξηγήσει και οι τροποποιήσεις που πρότεινε είναι εξαίρετες και μας επιτρέπουν καλύτερα να καταλάβουμε το θέμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν μιλάμε για την οδηγία που αφορά την ελάχιστη κατάρτιση που θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους ναυτικούς. Μιλάμε για την ε, μεταγραφή της σύμβασης S TCW που ήδη έχει υιοθετηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένα μέγα τμήμα τη οδηγία. αφορά άμεσα αυτή τη σύμβαση. Και άρα θα έπρεπε πραγματικά να προσέξουμε ε, ώστε να μην βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου δηλαδή η χώρες μέλη να πρέπει να υιοθετήσουν κείμενα, δύο κείμενα με διαφορές μεταξύ τους. Όσον αφορά τη σύμβαση, συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Κρίστενσεν ότι η μεταφορά, η διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα πιστοποιητικά και το επίπεδο των προσόντων των ναυτικών θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό της προστασίας των δεδομένων. Το σύστημα ενημέρωσης της σύμβασης STSW, το οποίο επεξεργάστηκε η, Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, είναι πάρα πολύ, ε, συγγνώμη, ο Διεθνής Ναυτιλικός Οργανισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, ε, είναι ζωτική σημασία για τις αγορές εργασία και μα επιτρέπει καλύτερα να προετοιμάσουμε τη σταδιοδρομία και την εργασία των ναυτικών. Θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με, με τις σχολές εκπαίδευσης των ναυτικών. Και όσον αφορά το περίοδο 18 μηνών, Πιστεύω πως οι κανόνες που ισχύουν σήμερα είναι πιο ρεαλιστικοί. Ο εισηγητής μίλησε επίσης για ώρες εργασίας και για ώρες ανάπαυσης. Και αυτά σε σχέση με την οδηγία που αφορά το χρόνο εργασίας. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Γνωρίζουμε πως σήμερα πολλά πλοία φέρουν σημαία άλλης χώρας, πράγμα το οποίο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Είναι δύσκολο να βρεθεί εδώ συμβιβαστική λύση, αλλά θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την οδηγία για την ελάχιστη εκπαίδευση των ναυτικών, πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία θα βελτιώσει την ασφάλεια στις θάλασσες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ήρσου. Thank you, Madam Chair. on behalf of our ALDE shadow, Philip... Εξ ονόματος του κυρίου Δεμπάκη, θα ήθελα να σας αναφέρω τις παρατηρήσεις του. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε για συνεργασία με τους διάφορους και εισηγητές, πράγμα που μας καθιστά πιο αποτελεσματικούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πολλής χώρο ε, ελιγμού όσον αφορά την μεταγραφή της Σύμβασης της Μανίλας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα, όπως ήδη αναφέρθηκε, πράγμα που καθιστά δύσκολη τροποποίηση του. Γι' αυτό πιστεύω πως η πρόταση Κομισιόν είναι καλή. Επίσης μπορώ να υποστηρίξω την άποψη του εισηγητή, συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις του και όσον αφορά την τροπολογία 24 για την προστασία των δεδομένων για την ομάδα μας και για την Άλντε, πολύ σημαντικό σημείο για... και μάλιστα ίσως θα υποβάλουμε πρόταση για ενίσχυση της. Ε, ίσως να έχουμε κάποια προβλήματα για το τροποποίηση του άρθρου 15 11, το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας ε, ίσως να είναι πρόβλημα και αν απαραίτητο θα υποβάλουμε σχετική τροπολογία. Οι τροπολογίες για την Συμφωνία της Μανίλα ήδη ξεκίνησαν, άρχισαν να ισχύουν στην 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και όσον αφορά την πρόταση της, της Κομισιόν χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Μπορεί να υπάρχουν ε, προβλήματα όσον αφορά τους λιμενικούς ελέγχους σε κράτη εκτός Ένωσης γιατί μπορεί κάποιες ε, να μην έχει εκδοθεί πιστοποίηση STCW του 2010. Έτσι μπορεί να σημειωθούν μεγαλύτερες ε, καθυστερήσεις, ε, τις οποίες θα πρέπει να δεχτούμε. Ωστόσο, πιστεύω πως η συμφωνία αυτή είναι απαραίτητη. Ολοκληρώνοντας, ε, να πω ότι υποστηρίζω την γνωμοδότηση, αλλά μπορεί να υποβάλω κάποιες τροπολογίες και προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκεώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανεί εξ ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Monsieur Mendola, au titre de la Commission. Thank you. Um, well, as mentioned... Ευχαριστώ. Όπως είπε η συγγήτρια, είναι πολύ τεχνικό Συγγήτρια. Ο εισηγητή, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ τεχνικό ε, το ζήτημα ε, και πρώτης, ε, πρώτη του 2012 είναι η ημερομηνία που έχει προβλεφθεί τον νέο κανονισμό. Καλωσορίζουμε την έκθεση. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Και όπως ακούσαμε και από τον κύριο Κρίστενσεν, ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ανάμεσα στο σετ κανόνων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύμβαση που ισχύει σε αυτό ε, το τομέα, η STCW δηλαδή. Ε, Ούτω ή άλλω αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε το περιεχόμενο τη σύμβαση STCW ε, στην κείμενη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω άλλα σχόλια. Σα ευχαριστούμε ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα βασιστώ σε αυτά για να καταλήξουμε σε ένα ευελπιστό εξισορροπημένο κείμενο. Όπως είπε ο κύριος Κοσλός και η κυρία Χίρσε για τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά, ε, αναφερόμαστε ήδη στο θέμα της προστασίας ε, των δεδομένων ε, και θα το έχουμε υπόψη μας ε, διότι Έχουν ενισχυθεί οι διατάξει ασφαλείας στην πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών. Χαίρομαι που ο κύριο Κοσλεύσκη αναφέρθηκε στην οδηγία για το χρόνο εργασία και το χρόνο ανάπαυσης. Θα προσθέσω αυτή τη διευκρίνηση στο κείμενο, διότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ερμηνεία των κανόνων. θα γινόταν όλη η διαδικασία πολύ περίπλοκη, αν δεν ίσχυε αυτό το κοινό σετ κανόνων. Ε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε θετικά για το σχέδιό μας. Βλέπω ότι είναι ευρία η συνένεση. Περιμένω τις τροπολογίες σας για να ρυθμίσω αυτά τα ζητήματα και όπως είπε ο κύριος Ντεπάκερ, ελπίζω και εγώ να καταλήξουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να συνεχίσουμε αυτή την τόσο καλή συνεργασία. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε. Η συνολική στρατηγική για να αποφύγετε τα θέματα φίλου είναι να τα λέτε στο πληθυντικό όλα. Καλό το σύστημα, μήπως να το εφαρμόσουμε γενικότερα. Ούτω ή άλλως ε, θα επανέλθουμε. Τελειώσαμε τώρα το σημείο 16. Και τώρα θα πάμε στο σημείο 10. Και θα δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρό μας, Κοινά διαχείριση. Για του 20 κύριου λόγου ανησυχία των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ε, λειτουργία τη ενιαία αγορά. Θα εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την ε, έκθεσή σας. 77 είναι αυτές. Änderungsanträge ähm, Σας ευχαριστώ πολύ. Hierfür und für οι περισσότερες τροπολογίες ε, έρχονται να συμπληρώσουν πολύ ωραία τη γνωμοδότησή μου ε, και ε, την εμπλουτίζουν με σημαντικά στοιχεία, τη βελτιώνουν. Ελπίζω να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε κάποιους συμβιβασμούς. Και ε, είναι λοιπόν ορισμένες τροπολογίες για την ίση αμοιβή που επί της ουσίας βρίσκω πολύ καλές και μπορώ απολύτως να συμφωνήσω. Ε, το ερώτημα βέβαια είναι Μήπως να το συζητήσουν ξανά οι σκιώδες ηγητές αν το θέμα της ίσης αμοιβή έχει χώρο εδώ. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό κάποιας μεμονωμένης χώρας, αφορά όλες τις χώρες. Δεν ξέρω, πραγματικά το λέω, αν επί της ουσίας ανήκει σε αυτή την έκθεση. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες οι οποίες θέτουν τις επιχειρήσεις υπό καθολική υποψία. Και υπονοεί ε, αυτό το σύνολο τροπολογιών ότι ε, ουσιαστικά η πλειονότητα των επιχειρήσεων εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε με μια τέτοια έκθεση αντιμέτωπους στους πολίτες με τις επιχειρήσεις. Ε, πάντως, την εβδομάδα του Στρασβούργου θα το ξανασυζητήσουμε και όλοι οι και εγώ, μήπως χρειαστεί να ξαναδούμε κάποια διατύπωση, να αναδιατυπώσουμε ορισμένε τροπολογίες. Κάτι άλλο που βρίσκω πολύ ωραίο είναι η ιδέα Ε, ενός 28ου συστήματος ε, ασφάλισης ε, και το ζητούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και μάλιστα δεν το προτείνουν εθελοντικά να ισχύσει αλλά από την αρχή υποχρεωτικά. Κοιτάξτε είναι πάρα πολύ τορμηρή ιδέα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δεχθούμε έτσι. δεν θα θέλατε σε μια πρώτη φάση να είναι εθελοντική, αλλιώς θα μπλέξουμε θα γίνουν πολλές ε, συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν πειράζει. Ας γίνει και αυτή η συζήτηση. Ένα άλλο σημείο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η τροπολογία υπαριθμών 17 που γίνεται λόγος εκεί για ένα κεντρικό σημείο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο σε περίπτωση που δεν υπάρχει, βεβαίω να το δημιουργήσουμε, να το προτείνουμε. Γιατί, Γιατί ο στάδιο της υλοποίησης είναι απολύτως απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προόδους και να συντονίζει οπωσδήποτε. Γιατί δεν είναι πάντα καλή η συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Αυτές οι ιδέες και με χαρά θα ακούσω τη συζήτηση με τους κοιόδους ηγητές και ελπίζω κάποια στιγμή και οι τροπολογίες αυτές, ορισμένες τουλάχιστον, να μπουν στην έκθεση και να ε, βρουν και τη συνένεση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόπε Φοντανιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια. Όντως υπάρχουν πολλά σημεία που εμείς θεωρούμε παρόμοιες τροπολογίες και πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω την εισηγήτρια. Έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου αν θα πρέπει να είναι το νέο σύστημα υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά για τις συντάξεις, την υγειονομική περίθελψη. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μετακινούμενους εργαζομένους, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά θα ήταν καλό να ε, το συζητήσουμε στο Στρασβούργο την εβδομάδα της Ολομέλειας. Πάντως ήδη ξέρει η συγκήτρια ότι το ΕΛΚ είναι στη διάθεσή της και μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Στάινμπουργκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 77 είναι οι τροπολογίες και σε μεγάλο βαθμό ε, πηγαίνουν σε σωστή κατεύθυνση και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό. Είμαι βέβαιη ότι θα γίνουν πολλές και εντατικές συζητήσεις σε μερικά σημεία γιατί οι βασικές αγωνίες των πολιτών είναι οι βασικές αγωνίες των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά. Δηλαδή και η αρχή της ίσης αμοιβή για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά όχι μόνο εμένα, το μεταφέρουν και σε άλλους αυτό. Επί της ουσίας τώρα για την κοινωνική ασφάλιση και προστασία των μετακινούμενων εργαζομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ως μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι ε, ένα τέτοιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που μπορεί κάποιος να ε, μεταφέρει τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί αυτό να είναι εθελοντικό ή προαιρετικό. Επίσης ενημέρωση για μετακινούμενους εργαζομένους. Το λέει αυτό παντού. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική ασφάλιση, αλλά θα πρέπει ε, να αφορά την ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ανέργων. Το θέμα του κεντρικού σημείου συντονισμού στα κράτη-μέλη το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ζήτησα στην τροπολογία μου 17 να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μου διαβιβάζουν πάρα πολλά προβλήματα που ανακύπτουν σε φορολογικό δίκαιο, στο ασφαλιστικό δίκαιο, στο εργατικό, στα μισθολογικά και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα λύσουν μόνοι τους αυτά και δεν τα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Εγώ ζω κοντά στα γαλλογερμανικά σύνορα και συναντώ πολλούς εργαζομένους που ζουν στην παραμεθόριο περιοχή και έχουν πραγματικά υπαρξιακά προβλήματα γιατί ισχύει διαφορετικό δίκαιο όταν δουλεύουν σε μια χώρα και κατοικούν στην άλλη. Ακόμα και αν είναι διμερείς συμφωνίες αυτές θα πρέπει να ειδωθούν σε κεντρικό επίπεδο. Μετά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που εισάγουν διακρίσεις. Το λένε και οι τροπολογίες ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των εργαζομένων ανδρών και γυναικών και εδώ είναι και θέμα τήρησης της ε, οδηγίας για την ίση μεταχείριση και ίση αμοιβή. Και δεν είναι μόνο εργαζόμενοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Για το θέμα της απόσπασης εργαζομένων ήρθαν κάποιες τροπολογίες από διάφορες κατεμβήσεις και πολιτικές ομάδες και έχει ιδιαίτερη σημασία η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να εγγυάται και η οδηγία αυτή ε, την ισότητα αμοιβών, να σέβεται τις συλλογικέ συμβάσεις και επίσης να μην ανοίγει το δρόμο για το κοινωνικό dumping. Αυτά. Εντάξει, 77 τροπολογίες έδειξαν ότι ο κόσμος εργάστηκε πολύ για την έκθεση. Αυτή είναι σημαντική. Αν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα, μάλλον το πόλιο αλλιώς θετικά. Εάν λύσουμε αυτά τα προβλήματα θα έχουμε τους πολίτες στο πλευρό μας και ε, θα ξεπεράσουμε αυτόν τον ανητισμό και την απαξίωση για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στη Ρεζίνα Μπάστος για να μας ε, ε, ε, εκφράσει την τοποθέτησή της ΣΥΝΚΟ θα ήθελα να σας πω κι εγώ κάποια πράγματα για τις εκθέσεις. Δεν έχω ε, υποβάλει τροπολογίες, βέβαια γι' αυτό εγώ φταίω, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η αντίληψη ή οι ανησυχίε ε, των Ευρωπαίων ότι μιλάμε για ιδιώτες και για επιχειρήσει ε, σε σχέση με την ενιαία αγορά. Περιορίζονται λοιπόν αυτέ οι ανησυχίε στη διασυνοριακή διάσταση του ζητήματο, αλλά δεν εξετάζεται καθόλου ο ρόλο της ενιαία αγοράς σε σχέση με τι εθνικέ πολιτικέ. Σας είχα μιλήσει παραδείγματο χάρη για τι εργατικέ κατοικίε, στην κοινωνική στέγη, ε, μια ιδιαίτερα επίκαιρη ιδέα, εφόσον συζητούμε και τον ανταγωνισμό γιατι γιατί κάποια κράτη-μέλη ίσως ε, δεν δίνεται να αναπτύξουν αυτόνομες ε, εθνικές πολιτικές ε, κοινωνικής και εργατική στέγης λόγω της έλλειψης συντονισμού. Δεν έχω υποβάλει τροπολογίες και ξαναλέω είναι δικό μου το λάθος, αλλά έτσι είναι. Η κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και να της ευχηθώ καλή επιτυχία για τις ε, τροπολογίες. Ε, καλή τύχη γιατί υπάρχουν 77 τροπολογίες, ε, πάρα πολλές και αυτή η έκθεση θα είναι μία από τις 7 εκθέσεις που θα ενοποιηθούν σε ένα συνολικό κείμενο για το οποίο είμαι εγώ εισηγήτρια εξ ονόματος Επιτροπής ΙΜΚΟ. όλοι θέλουν να είναι εστιασμένη και συνεκτική η έκθεση, ε, κυρίως επειδή έχει αυτό τον απότερο στόχο να ενταχθεί σε μια συνολικότερη έκθεση. Χρειάζεται λοιπόν ε, η απαιτούμενη εστίαση σε αυτά τα 20 προβλήματα που παρατηρούνται ε, στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ήδη έχουν ξεκαθαριστεί οι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Απασχόληση σε σχέση με τι 20 βασικέ αυτέ ανησυχίε. Επειδή είμαι εισηγήτρια στην Βασική Επιτροπή, ήθελα να το τονίσω ακόμη περισσότερο. Ε, το θέμα της ε, ε, κοινωνικής ασφάλισης, απαραίτητο για τους εργαζομένους, η ατροφαρμακευτική περίθαλψη, άλλο εκ των ονουκάνευ, κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης, όλα αυτά τα ζητήματα είναι της αρμοδιότητάς σας και γνωρίζουμε ότι θα είναι μια σημαντική συμβολή στην τελική έκθεση. Επίσης θα πρέπει να διαφαίνεται ήδη ο στόχος της τελικής έκθεσης έκθεσης. Ε, δηλαδή να μην ζητούμε με μονομένες λύσεις, 20 διαφορετικές λύσεις για τις 20 διαφορετικές ανησυχίες δηλαδή, αντιπροτείνουμε να εκπονήσουμε τις βασικότερες ε, συστάσεις ούτως ώστε και ε, η Ένωση και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση σε αυτές τις 20 ανησυχίες. Τρία είναι τα βασικά κεφάλαια. Πρώτον, ενημέρωση των ε, ε, πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα ε, προνόμια και τα δικαιώματα που έχουν μέσα στην εσωτερική αγορά, γιατί η εσωτερική αγορά είναι αυτή που φτιάχνει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Δεύτερον, μεταφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, γιατί ορισμένες φορές δεν γίνεται αυτό σχολαστικά από τα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί σωστά όχι η διεθνή νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία διορθώνει ομιλήτρια και έτσι να εξασφαλίσουμε σε εθνικό επίπεδο καλύτερη διακυβέρνηση. Συνοψίζω. Με την ιδιότητα της εισηγήτριας, αυτή είναι η βασική μου ανησυχία, να περάσει το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση, αφοσίωση και κυρίως πολιτική βούληση ώστε να άρουμε αυτούς τους ε, φραγμούς παρακολύουν την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τρόπο ώστε ε, σε αυτή την περίοδο της κρίσης σε αυτή την περίοδο μεγάλου σκεπτικισμού σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες ε, και πάλι να καταφέρουν να πάρουν αυτό το μήνυμα ελπίδας, αλλά όχι μέσω μόνο της άρσης των φραγμών που τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας ενιαίας αγοράς εξακολουθούν να υπάρχουν. Ξαναλέω ότι θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας μέσα στην έκθεση σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που ήδη έχουμε συζητήσει, όπως είπε και η συνάδελφος ε, η Βερόνικα για τα στήματα αρμοδιότητας της ΕΙΜΚΟ, ιατροφαρμακευτική φαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή κινητικότητα κτλ. Να υπάρχει κατάλληλη εστίαση μέσα στην έκθεση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο, οπότε θα ξανακούσουμε την κυρία Χίρσο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας ε, ως απάντηση στα όσα είπα. Βεβαίως θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε κάποιες μικρές ε, εξουσίες εδώ και αρμοδιότητες και θα πρέπει να φαίνονται στην γνωμοδότηση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στο συμβιβαστικών τροπολογιών και θα προσπαθήσουμε τις ερχόμενες εβδομάδες να το συζητήσουμε σε συνεργασία με τους εκάστοτε συντάκτες των τροπολογιών έτσι ώστε στο Στρασβούργο να είμαστε έτοιμοι και να προκάνουμε. Ελπίζω να συμφωνήσουμε για τα περισσότερα και να στείλουμε στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ένα σαφές μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, η Πρόεδρος. Λοιπόν, Κατόπιν τούτου θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας, δηλαδή 23 και 24 Απριλίου. Θα έχετε κάνει μέχρι τότε τις συμβαστικές τροπολογίες ή όχι. Ε, τότε στις 23 θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και στις 24 θα ψηφίσουμε για να μπορέσει και η Επιτροπή ΙΜΚΟ εσωτερικής αγοράς να το κοιτάξει, που είναι καθέλη αρμόδια, με εισηγήτρια την κυρία Μπαστός. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 18. Ο κύριος Κόζα απουσιάζει. Α, το έχει αναλάβει άλλο συνάδελφος το θέμα του. Ε, πρόσωπος του κυρίου Κόζα. Ο κύριος Σούζα. Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017, εξέταση σχεδίου γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο. Thank <coughs> Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κούσα δεν μπορούσε να είναι παρόν, γι' αυτό και μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή του. Θα τη διαβάσω στα ουγγρικά. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα ανάμεσα στο 1900, το 2013 και το 2019 είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα γιατί αυξάνεται η ζήτηση, συγγνώμη, 2013-2017 ε, είναι πολύ φιλόδοξο γιατί ευκράνεται η ζήτηση για περισσότερες και ακριβέστερες στατιστικές. Το ίδιο ηθεί και τον ευρωπαϊκό ε, χώρο, τα στοιχεία αυτά τα χρειαζόμαστε γρήγορα και πρέπει να μπορούν και να ερμηνευθούν πιο εύκολα, καθώς και να είναι και πιο προσβάσιμα. Φυσικά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι τα μέτρα λιτότητας ε, καθιστούν δύσκολη την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Το νέο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα είναι απαραίτητο έτσι ώστε οι στατιστικολόγοι να μιλάνε με τα ίδια στατιστικά στοιχεία και να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες το κάθε κράτος μελος Χρειάζεται πραγματική συνεργασία ανάμεσα στο, στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και ε, μάλιστα συνεργασία επαγγελματικού τύπου έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να τονίσω την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα στατιστικά αυτά στοιχεία. Η πρόεδρος ε, ειδοποιεί τον ε, ομιλητή να μιλά λίγο πιο αργά. Μιλάμε επίσης για νέους δείκτες. Όταν ε, μιλάμε για νέους δείκτες θα πρέπει να βασιζόμαστε στι φυστάμενες στατιστικές και πληροφορίες. Πέρα από τους δείκτες για την ανάπτυξη, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται δείκτες για την παραγωγικότητα. Υπάρχουν άλλοι δείκτες οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη και έπειτα υπάρχουν διάφορες ιδέες και στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούν αν θέλουμε τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν να είναι σε θέση να προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της εξελίξης θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, χρήση των ε, σχετικών δικτών ώστε να λάβουμε υπόψη ότι αν θέλουμε να είναι διαθέσιμοι οι δημόσιοι χώροι για άτομα με ειδικές ανάγκες, χρειαζόμαστε και τις κατάλληλες στατιστικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προγραμματίζει να δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την πρόσβαση στους δημόσιους χώρους και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την γύρανση του πληθυσμού καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό και η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Κοινωνική πρόνοια, υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ε, προτεραιότητα για μια βιώσιμη κοινωνία. Τώρα όσον αφορά τις μεταφορές χρειαζόμαστε στατιστικές που να δείχνουν το επίπεδο προσβασιμότητας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου στατιστικέ για το ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικέ ανάγκε όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα μεταφορά. Και κατά πόσο τα μέσα αυτά είναι προσαρμοσμένα ε, στα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω ανάπτυξη δικτών σε αυτό το επίπεδο, σε ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτές οι στατιστικές θα πρέπει να είναι και φιλικές προς τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ, ο κύριος Μπένιον. Μάλιστα. Εν γέννη νομίζω πως οι περισσότερες ε, τροπολογίες προσφέρουν κάτι νέο, το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την χρήση του λέξης barrier free, ανεφραγμών, στην ε, τροπολογία 10 και 9 χωρίς φραγμούς είναι κάτι το πολύ απόλυτο. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε την φράση άνευ περιορισμών. Μιλάμε δηλαδή για constraints on accessibility. Περιορισμοί της πρόσβασης. Ε, σημαίνει αυτό ότι διαρκώς υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ακόμα και αυτοί που είμαστε και ρεοί σωματικά και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, δεν, είμαστε, ε, δεν έχουμε πρόσβαση χωρίς φραγμούς. Ας πούμε οι νέοι δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο γιατί δεν έχουν τα χρήματα να τα αγοράσουν και να, γιατί δεν έχουν δίπλωμα κτλ. κτλ. Είναι πολύ απόλυτη αυτή η φράση ανεφραγμών φραγμών, χωρίς φραγμούς ε, στα ελληνικά, το barrier free Τροπολογία 5. Στηρίζω την άποψη ότι θα πρέπει οι νέοι δείκτες όσο είναι δυνατόν ε, να βασίζονται στα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για δύο βασικούς λόγους. Δεν είναι μόνο το κόστος που είναι βέβαια ένας από τους λόγους, αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι σημαίνει ότι αν κανείς αντλήσει στοιχεία από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, σημαίνει πως έχει στη διάθεσή του έτσι και ιστορικά στοιχεία και άρα μπορεί να βγάλει τις τάσεις άμεσα. Ενώ αν ξεκινήσει με νέα σύνολα στοιχείων, όχι μόνο κοστίζει περισσότερο, αλλά και για 5, 6, 7 χρόνια δεν θα μπορεί να, έχει, να, να, να εξετάσει τάσεις. Εκεί όπου είναι δυνατόν λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Η τροπολογία 6 δεν με πείθει όσον αφορά την αφαίρεση της παραγωγικότητας, θα το σκεφτώ δεν ξέρω κατά πόσο περιτεύει. Εγώ σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να έχουμε στοιχεία για την παραγωγικότητα και θα πρέπει να με πείσετε για αυτήν. Και για την τροπολογία 13 νομίζω ότι ε, χρησιμοποιεί μια γλώσσα που είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφήσει κανείς ενώ η αρχική διατύπωση είναι πιο εύληπτη και θα την προτιμήσω. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει τον λόγο. Εγώ μέσω του κυρίου Σόγκορ θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κόζα να σκεφτεί ποια είναι η ισορροπία του προγράμματος που προτείνεται εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί φαντάζομαι πως αυτό το στατιστικό πρόγραμμα έρχεται για να στηρίξει πολλές πολιτικές που ξεκινούν ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σκεφτούμε πούμε όλο το θέμα της ε, μακροοικονομικής εκτέλεσης, της οικονομίας ή την στρατηγική Ευρωπαϊκή 2020 και την επίτευξη των στόχων της, ε, των στόχο καταπολέμησης της φτώχειας, είναι αλήθεια ότι σε αυτό το τομέα έχουμε ένα πρόβλημα συλλογής πληροφοριών φρικτό. Δηλαδή, σοβούς της κρίσης των subprime είχαμε ως ενημέρωση την πιο πρόσφατη μάλλον ενημέρωση που είχαμε, οι πληροφορίες που είχαμε, δίναν ε, την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία χρόνια πριν. Οι τροπολογίες λοιπόν είναι σημαντικές, αλλά πέρα από αυτές δεν είχα βέβαια και την ευκαιρία να δω όλες τις λεπτομέρειες. Ανησυχώ λοιπόν, μήπως τελικά εμείς ξεκινάμε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ισορροπημένο τρόπο. Και αν οι δείκτες για τους οποίους ας πούμε η Βελγική Προεδρία έχει πολύ εργαστεί, λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το πρόγραμμα στατιστικών. Δεν υπάρχει εδώ κάποιος από την Κομισιόν. Α, υπάρχει. Μάλιστα. Ίσως λοιπόν από πλευρά της Κομισιόν θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτές τις ε, ανησυχίες, προβληματισμούς για να δούμε μετά πώς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε επί της ουσίας. Λυπούμε αλλά δεν έχω το όνομά σας, οπότε αν γίνεται ε, να μας το πείτε πριν απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Γιλιέρμο Ντάβιλα και αντικαθιστώ τον υπεύθυνο συνάδελφο που είναι αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο και δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι παρόν στη σημερινή συζήτηση. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Πρόεδρο ε, για την, την γνωμοδότηση αυτή που έχει ετοιμάσει αυτή την Επιτροπή λαμβάνουμε υπόψη, μάλλον σημειώνουμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και συζητήθηκαν σήμερα. Θεωρούμε πως είναι θεμητές και ε, τις μελετούμε. Μια σύντομη αντίδραση στις δικές σας παρατηρήσεις σήμερα, καταρχήν όσον αφορά το θέμα της ανταγωνιστικότητας, τα στοιχεία δηλαδή, τη βάση δεδομένων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Κόζακ ότι ακριβώς αυτός ο τίτλος καλύπτει δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν και που λειτουργούν και μέσα στο πλαίσιο των στατιστικού προγράμματος αναπτύσσουμε στατιστικές που στηρίζουν αυτή την ανάλυση. Δεν ζητάμε νέες πρωτοβουλίες, απλώς θέλουμε να δώσουμε νομική βάση στις, ε, στις προτεραιότητες που ήδη ε, κάνουμε σε αυτό το τομέα. Η τροπολογία 6 λοιπόν ίσως να μην είναι σκόπιμη. Και όσον αφορά το θέμα της κατάρτισης και της προσβασιμότητας για τους πολίτες, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σας ότι εδώ θέλουμε να εισάγουμε αυτή την ιδέα ότι όχι μόνο μιλάμε για την κατάρτιση των χρηστών, αλλά των πολιτών ευρύτερα, πέρα δηλαδή από τα μέσα της... Ε, αποκλειστικά της Κομισιόν. Θέλουμε φυσικά ε, η πρόσβαση και η κατανόηση για τα στοιχεία μας να είναι όσο γίνεται καλύτερη. Επίσης, όσον αφορά τους δείκτες για το 2020 ε, και για την διευκρίνηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, φυσικά ε, θεωρούμε και είδατε τον πρώτο πίνακα επιδόσεων, ε, θεωρούμε ότι έχουμε πολύ στέρεες συμπαγής βάσεις για τις στατιστικές μας. Εργαζόμαστε για τη βελτίωσή τους. Είναι ένα παραδοσιακό πρόβλημα που έχουμε ωστόσο, ότι είναι λιγότερο ταχεία η απόδοσή μας όσον αφορά τις στατιστικές για την ανεργία προσπαθούμε να βελτιωθούμε και χρησιμοποιούμε και ένα νέο όραμα για το πώς να εξυγχρονίσουμε τις ε, μεθόδους παραγωγής στη στατιστική εργασία, πράγμα που πρόθεσμα θα μας βοηθήσει, ώστε αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα και για τον τομέα της ε, απασχόλησης. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος εισηγητής, θέλετε να παρέμβετε, κύριος Σογκόρ. όχι κοιτάξτε να διαβιβάσετε πιστά τη συζήτηση στον εισηγητή μας. Έχουμε λοιπόν προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 4 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και θα εξεταστούν στην συνεδρία στις 23 και 24 Απριλίου. Θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές στις 30 Μαΐου για να τις ψηφίσουμε στις 31. Η ΕΚΟΝ θα ψηφίσει στις 18 Ιουνίου το θέμα αυτό. Και τελευταίο σημείο της σημερινής ε, των εργασιών μας είναι η πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας σε σχέση με το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλασφάλισης για το οποίο θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μπάστος. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο Είμαστε σε διαδικασία συνδεδεμένη επιτροπή με την νομική επιτροπή και επί τη οποία η οικονομική και νομισματική επιτροπή θα γνωμοδοτήσει. Κυρία Εισηγήτρια, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Αυτό το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλασφάλισης είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Ήμασταν η αρμόδια επιτροπή σε πρώτο στάδιο για την βασική έκθεση και στη συνέχεια η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων διεκδίκησε ε, την βασική αρμοδιότητα για αυτό το ζήτημα και εμείς ε, ε, λοιπόν είμαστε συνδεδεμένη επιτροπή πλέον. Αυτό μας περιορίζει κατά τι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από πλευρά τη Επιτροπή μα. Έφτασε η στιγμή να αναλυθεί η νομοθετική πρωτοβουλία για ένα καταστατικό των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλασφάλισης το 92, εδώ και 20 χρόνια έχει αυτή η διαδικασία, από το 92 ζητά αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία το Κοινοβούλιο και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει σχέδιο κανονισμού, το οποίο όμως το 2006 τελικά αποσύρθηκε από την Επιτροπή και λυπούμαστε γι' αυτό. το κεντρικό ε, σημείο, αν θέλετε, το της έκθεσης είναι να έχουν νομικά μέσα στη διάθεσή τους αυτά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλασφάλισης, ε, τα οποία θα διευκολύνουν την ε, λειτουργία τους στην εσωτερική αγορά, δηλαδή σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια μεγάλη παράδοση σε ταμεία αλληλασφάλισης. Σε άλλα κράτη δεν υπάρχουν τέτοια ταμεία. Ε, μπορώ και να κατονομήσω, κατονομάσω αυτές τις χώρες. Εστονία, Τσεχία, Λιθουανία και Σλοβακία. Δεν υπάρχει καν ταμείο αλληλασφάλισης. Αντίθετα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες υπάρχει μια πολύ μακρά παράδοση αυτών των ταμείων σε κάθε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι είναι τόσο βαθιά ριζωμένη αυτή η παράδοση σε κάποιες κοινωνίες ώστε ε, μπορεί να θεωρηθούν τα ταμεία αλληλασφάλισης ως ένα συμπλήρωμα του κράτους πρόνοιας ή και του ε, κοινωνικού προτύπου, του προτύπου κοινωνικής ασφάλισης, της προστασίας, της υγείας των κρατών μέλων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτών των ταμείων και γι' αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα αυτά τα μία ε, νομίζω δικαιούνται μία απλούστευση ως προς τη λειτουργία τους μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον κυρίως κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όπου τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ε, τα εθνικά συστήματα υγείας παραπέουν και δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουν από χρηματοοικονομικής ε, πλευράς. Ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνική προστασία, ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνική ασφάλεια διενεργείται μέσω αυτών των ταμείων αλληλασφάλιση ε, και άρα χρειάζονται συγκεκριμένα εργαλεία στη διάθεσή του, ούτω ώστε να μπορέσουν να δράσουν επί ε, μία ε, βασιζόμενη σε μία κοινή πλατφόρμα, αν θέλει, σε μία κοινή δέσμη κανόνων που θα ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, τα ταμεία αλληλασφάλισης ασφαλίζουν περίπου 160 εκατομμύρια ανθρώπους ε, στην ε, Ένωση και βοηθούν ε, και την απασχόληση, διότι απασχολούν 350.000 ε, ανθρώπους. 20% ε, της αγοράς ασφαλείων κατέχουν και μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων ασφαλιστικών δηλαδή εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το ειδικό τους βάρος μέσα στην εσωτερική αγορά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοούμε πια αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε το, ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο ε, των συστάσεών μας και να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι ούτω ώστε να παρακινήσουμε την Επιτροπή ε, για να εισηγηθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ακολουθήσει τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία στη συνέχεια χάρη στην οποία θα λειτουργούν πιο εύρυθμα αυτά τα ταμεία ασφάλισης μέσα στην εσωτερική αγορά. Περιμένω λοιπόν τις ε, παρατηρήσεις και τις τροπολογίες ε, των σχεδόν εισηγητών και όλων των συναδέλφων και επιτρέψτε μου Πρόεδρε να σας μιλήσω λίγο για το χρονοδιάγραμμα ήδη τώρα. τόσο για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όσο και για τη δική μας. Ε, στις 10 Απριλίου μέχρι τις 12 ε, είναι η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Στη συνέχεια εξέταση των τροπολογιών 30 και 31 Μαΐου και κατόπιν συμβαστικές τροπολογίες και έγκριση της έκθεσης στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. Ενώ στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων η πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρίς έγγραφο ε, θα γίνει στις 18 ε, και 19 Ιουνίου και η εξέταση της έκθεσης θα γίνει στις 9 ή στις 10 Ιουλίου μετά ο 11 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία για τι ε, πρωτοβουλίε και 10-11 Οκτωβρίου θα εξεταστούν αυτέ τι τροπολογίες. Κατόπιν θα εγκριθεί στην Βασική Επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων αυτή η έκθεση τον Νοέμβριο. Ε, είναι καλό να έχουμε το χρονοδιάγραμμα κατά νου για να εργαστούμε για αυτό το συμβολική σημασία ζήτημα στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Euh, Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκεν. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω πόσο σημαντικό για μας ε, τους σοσιαλδημοκράτες είναι αυτό το θέμα, όχι μόνο τα ταμεία ελασφάλισης, αλλά και το ευρωπαϊκό καθεστώς για αυτές τις εταιρείες. Γιατί με την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους, το δημοκρατικό τρόπο λειτουργία τους και ακριβώς το μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα είναι σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας. Και με το ευρωπαϊκό καθεστώς αυτές οι ε, μορφές ε, εταιριών που παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές ε, χώρες θα έχουν την ευκαιρία να λειτουργούν πλέον και διασυνοριακά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, το είπε και η συγγήτρια άλλωστε, διότι πολλοί άνθρωποι δραστηριοποιούνται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε το σημείο 6, γιατί μπορεί να συμφωνώ με την άποψη ότι ενδεχομένως τα κράτη-μέλη να μπορούσαν να εμφανίζουν την ένταση ή την τάση μάλλον να μειώνουν τη δική τους συνεισφορά στην κοινωνική ασφάλιση. Αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αντισταθμιστεί από τα ταμεία ασφάλισης. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις δικές τους κοινωνικές ευθύνε και τις εισφορές τους και τα υπόλοιπα σημεία είναι, ε, συστήματα μάλλον να είναι απλώς επικουρικά της βασικής σύνταξης. Ε, ήθελα να ξαναστηρίσουμε και το 12 στη γερμανική μετάφραση γίνεται λόγος για την καταχώρησή τους σε κάποιο μητρό, αλλά δεν κάνουν ε, κέρδη. Δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, απλώς θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο οικονομικά αποδοτικό για να μπορούν να επανεπενδύουν στη δραστηριότητά τους. Αυτό άλλωστε είναι και η ιδιαιτερότητα αλλά και η ισχύ τους. Γι' αυτό το λόγο εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουμε ε, αυτή την κατάσταση και θα απορρίψουμε ό,τι απέχει και αφήσατε από την ε, υπόθεση της Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε με τις προθεσμίες. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού είμαστε συνδεδεμένη επιτροπή. Και τώρα πώς έχει η κατάσταση. Η έκθεση της Επιτροπής ε, νομικών υποθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα και το θεωρώ προβληματικό να πρέπει εμείς να εγκρίνουμε τη γνωμοδότησή μας χωρίς να έχουμε την έκθεση. Διότι μπορεί να είναι με ένα έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά είναι έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας. Καλό θα ήταν να έχουμε την έκθεση για να μπορέσουμε στοχευμένα να παρέμβουμε ε, με τροπολογίες να πάρουμε θέση. Θα σας παρακαλούσα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Έχουμε όντως τη δυνατότητα ή δεν την έχουμε ε, να κάνουμε τροπολογίες με το λόγο γνώσεως, δηλαδή να μας έχει έρθει η έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Μπάστος για την γνωμοδότησή της. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να Έχω καθυστερήσει ε, λίγο να ασχοληθώ με αυτό το τομέα σε σχέση με άλλους συναδελφούς, αλλά έχω μεγάλο θαυμασμό για τις εταιρείες αυτές και εδώ και καιρό ε, πιέζουν ε, να υπάρξει ένα καθεστώς. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία της πρόταση και ήθελα να ρωτήσω, ξέρω ότι το πρόβλημα είναι με το Συμβούλιο και αν σφάλω διορθώστε με. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, έκτοτε έχει αλλάξει τίποτα πήραμε κανένα δίδαγμα, ας πούμε για το καθεστώς των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών που να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκα αυτά τα θέματα και ανησυχώ γιατί θέλω να βοηθήσουμε με αυτά που θα κάνουμε και όχι να τους εμποδίσουμε. Ξέρω και πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ελλασφάλισης, αλλά θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ε, έχουμε τελικά ε, ανεπιθύμητες συνέπειες. Γι' αυτό ερωτώ, τι μαθήματα έχουμε μάθει από ε, τους συνεταιρισμού, από άλλα αντίστοιχα θέματα και ότι όταν λειτουργεί κάτι να λειτουργεί σωστά. Στη χώρα μου, τα, οι βασικότερες μορφές ανασφάλισης είναι τα Και ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε αντίθεση με τις τράπεζες δεν χρειάστηκαν διάσωση με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Ε, ήταν εύρωστες επιχειρήσεις και βλέπετε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια και μέσα φερεγγιότητας ε, και για οργανισμούς, Ινστιτούτα που αντλούν τους πόρους από τα μέλη τους είναι δύσκολο να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσει φερεγγιότητας στο ύψος του κεφαλαίου που χρειάζεται ε, να ασκούν το έργο τους και να ανταγωνίζονται παράλληλα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γι' αυτό ερωτώ. Δεν έχω καθόλου υπόψη μου ποια είναι η απάντηση. θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Ε, τα, τα μύρια ασφάλισης λοιπόν ε, είναι και πιο κρατεά και πιο αηφόρα. Γι' αυτό θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Επανέρχομαι όμως αυτό που είπα προηγουμένως. Έχω πλήρη επίγνωση ότι ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι βοηθάει παρά εμποδίζει. Σίγουρα προσωπικά δεν πρόκειται να υποστηρίξω τίποτα που να ε, πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, να ε, αποδυναμώνει την αλληλασφάλιση. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα πλέον ε, νομολογίας ε, του ΔΕΚ για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις που να μπορούμε να συμβουλευτούμε για να διδαχθούμε και από αυτές. Ευχαριστώ και προβλέπω στην συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους και εισηγητές και ελπίζω τελικά να είναι πολύ χρήσιμη αυτή μας η γνωμοδότηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και αυτό που είπε η κυρία Χάρκιν για τα διδάγματα που αντλήσαμε στην Επιτροπή μας όταν εκρίναμε την έκθεση Giggold για το ε, απολογισμό του καθεστώτος των συνεταιρισμών είναι πολύ σημαντικά. Γιατί αυτό το καθεστώς λίγο μόνο έχει χρησιμοποιηθεί προς το παρόν. Και κρίμα να μην βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επηρεάζει τελικά ε, το τοπίο και την αρχιτεκτονική ε, και τη λειτουργία των φορέων σε τομείς που δραστηριοποιούνται αυτά τα ταμεία ελασφάλισης. Τα γνωρίζω αυτά και ακριβώς μετά την απόσταση της πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, με τη δικαιολογία ότι είχε υπάρξει εμπλοκή, τα ταμεία ελασφάλισης προσπάθησαν να συνεργαστούν για να δουν πώς θα καταρτήσουν ένα στοιχειώδες ευρωπαϊκό καθεστώς. Ίσως πριν αποφανθούμε για την έκθεσή σας, καλό θα ήταν να κάνουμε και μία ακρόαση, αν θέλετε, με κάποια από αυτά τα ταμεία ελασφάλιση αλλά κατάλαβα ότι θέλετε να ακολουθήσετε ένα χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ σφιχτό και επιταχυμένο. Γιατί εμείς θα πρέπει να καλπάσουμε ε, και να οδηγούμε την κούρσα ενώ η νομική επιτροπή ε, καθυστερεί. Ε, βλέπω εδώ 6 Νοεμβρίου να λέει Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να καταθέσει μια πρωτοβουλία τέλη του έτους. Δεν ξέρω ασφάλω μπορείτε να με διορθώσετε για το στοιχείο αυτό του χρονοδιαγράμματος. Τι μορφή θα πάρει η πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την πρωτοπορία που έχουμε και τη χρονική άνεση, γιατί κάναμε και μια μελέτη, αναθέσαμε μια μελέτη ποιοτική. Γιατί αν θέλουμε εμείς να τρέξουμε υπερβολικά, ενδεχομένως να επιβάλλουμε στα ταμεία πράγματα που δεν θέλουν. Δεν μπορεί κάποιος έξωθεν να έρχεται να σας επιβάλλει. Εγώ δεν μιλώ για κανένα κράτος συγκεκριμένα της Ένωσης, έτσι το είπα. Ε, δεν είναι λοιπόν πάντα το πιο αποτελεσματικό κάποιοι άλλοι να σου λένε τι να κάνεις. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με την ακρόαση για να δούμε αυτά και τα χρονικά. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δικές πρωτοβουλίες να μας πει πού είναι τα πράγματα. Και τον τύπο και την ουσία και το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως η Κομισιόν από τον Οκτώβριο θέλησε να χρηματοδοτήσει μία μελέτη που ήδη προβλεπόταν από την ανακοίνωση σε σχέση με την πρωτοβουλία για την ε, πρωτοβουλία κοινωνικών ε, ε, επιχειρήσεων, Social Business Initiative, έτσι ώστε να δει ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση για τις εταιρείες αλληλασφάλισης στην Ευρώπη. Πρόκειται για την εξέταση όλων των εμποδίων όπου πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συνεταιρισμοί όταν θέλουν να επεκταθούν πέραν των συνόρων τους. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένονται για τα τέλη του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οπότε δεν ξέρω αν το χρονοδιάγραμμά σας συμπίπτει με το δικό μας, αλλά θα ήταν καλό να λάβετε υπόψη αυτή την ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να τονίσω ότι η ιδέα του κανονισμού αυτού είναι ιδιαίτερα προσφυλή στην Κομισιόν φυσικά, αλλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης που έγινε στο Συμβούλιο σε σχέση με την πρόταση κανονισμού στις αρχές του, της δεκαετίας του 90, αντιμετωπίσαμε προβλήματα, διότι όπως αναφέρεται στην έκθεση, η νομική μορφή των των Ταμείων Αλληλασφάλιση δεν, δεν υπήρχε σε όλα τα κράτη-μέλη, πράγμα που δημιουργούσε μια επιπλέον δυσκολία όσον αφορά τι διαπραγματεύσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη φυσικά τα εχθνά αποτελέσματα σε σχέση με την χρήση του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού. Είχαμε μόνο 24 Ευρωπαϊκούς Συνεταιρισμού μέχρι σήμερα και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης ε, που έκανε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, ε, την ξεκίνησε το περισμένο μήνα, σε σχέση με το μέλλον των ε, δικαιωμάτων των του εταιρικού δικαίου. Και, αυτό, και εκεί ένα από τα θέματα είναι ε, η σκοπιμότητα και η ανάγκη μιας τέτοιας, ε, ε, τέτοιων καθεστώτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μας, δεν προβλέπεται καμία σχετική κίνηση από πλευρά τη Κομισιόν μέχρι ότου ολοκληρωθούν αυτές οι δράσεις, η μελέτη δηλαδή και η δημόσια διαβούλευση. Βεβαίως υπάρχει επίσης η πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος που βρίσκεται τώρα ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η υποδοχή που θα τις επιφυλάξουν τα κράτη-μέλη, διότι θα ήθελα να τονίσω ότι όταν η Κομισιόν ε, αποφάσισε το 2006 να αποσύρει την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλασφάλισης και για την Ευρωπαϊκή ε, το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο, μόνο δύο κράτη-μέλη, το Βέλγιο και η Γαλλία, αντιτάχθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι συμφώνησαν. Και φυσικά τονίζω ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί θα πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα. Αυτό είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οπότε καταλαβαίνετε ποιες δυσκολίες προκύπτουν. Δεν είναι στο επίπεδο της Κομισιόν που μπορεί να κάνει την πρόταση, αλλά που δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο Συμβουλίου. Να σας πω ότι η πρωτοβουλία για το κοινωνικό επιχειρήν προβλέπει μια μελέτη για την ε, διατήρηση των ταμείων αλληλασφάλισης σε περίπτωση μετατροπής των ταμείων αλληλασφάλισης όπως έγινε στην Βρετανία πριν από 15 χρόνια περίπου της μετατροπής αυτών των ταμείων σε ανώνυμες εταιρείε. Η ιδέα είναι να δούμε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την προστασία του κληροδοτήματος που έχει συγκεντρωθεί για χρόνια να προστατευτούν δηλαδή τα ταμεία αυτά από την απώλεια της, ε, του κληροδοτήματός τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, το να αναλαμβάνει το δικαίωμα πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετικό είναι, αλλά ο στόχος, ξέρετε, ήταν ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη μελέτη που ε, χρηματοδοτήσαμε εμείς, πέρα από τη μελέτη και τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχει το δικαίωμα λοιπόν το Κοινοβούλιο να τροφοδοτεί τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν καταλήξουν στην τελική πρόταση που θα καταθέσουν ο στόχος να φτάσει στην Ολομέλεια αυτό το θέμα πριν το πέρας ε, του τρέχοντος ε, ε, μου φαίνεται ρεαλιστικός στόχος. Θα ρωτήσω την εισηγήτρια μας μήπως θα μπορούσαμε να παρατείνουμε την περίοδο που έχουμε στη διάθεσή μας για την υποβολή τροπολογιών για να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και να εξετάσουμε εκ του το θέμα. Να παρατείνουμε λοιπόν αυτή την ε, ε, προθεσμία και να τις προτείνω επίσης να διοργανωθεί μια ακρόαση για το καθεστώς ε, των Ταμείων Αλληλασφάλισης, ούτως ώστε τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, δηλαδή υγεία και κοινωνική προστασία, στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας, μέσα σε αυτή την ακρόαση να ακούσουμε ανθρώπους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον ή και ειδικού που θα μας ενημερώσουν για το καθεστώς αυτών των ταμείων, όπως μας μας είπατε κι εσείς, ε, σε κάποια κράτη δεν υπάρχει καν ε, τέτοιο ταμείο αλληλασφάλισης. Έχουμε και σχετική νομολογία του 10 κτλ. Τι λέτε κυρία Μπάστος, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις Σίμπουρ και Χάρκιν για τις για τη συμβολή τους σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομικό καθεστώς καθώς και την μελέτη και τη διαβούλευση που κάνουμε για το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα Ταμεία Αλληλασφάλισης. Τώρα, ως προς το συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτών των Ταμείων Αλληλασφάλισης, συμπληρωματικό ενώντας σε σχέση με τα εθνικά συστήματα, ε, θέλουμε να το αναφέρουμε χωρίς όμως να διαγράψουμε την αναφορά και να μην αναγνωρίζουμε τη σημασία των εθνικών συστημάτων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης ε, που είναι καθοριστική σε εθνικό επίπεδο. ως προς ε, την βιωσιμότητα αυτών των συστημάτων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλατήσκαλο ευρωπαϊκό κοινών ε, αξιών, μια βάση για να αναπτυχθεί μελλοντικά το καθεστώς ε, με στόχο, ναι μεν την κερδοφορία, αλλά όχι μόνο. Και εξάλλου η κερδοφορία δεν είναι αρνητική έννοια, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι όμως ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος είναι η επιστροφή των εισφορών στους ασφαλισμένους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να τονιστεί επαρκώς. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι, συγκεκριμένα η συνάδελφος Χαρκίν, θα πρέπει να ε, έχουμε όλες τις δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή να με την έκθεσή μας ε, να προκαλέσουμε, αν θέλετε, μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να καλύψουμε αυτό το ιστορικό κενό, διότι τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ διεκδικούν ένα ενιαίο καθεστώς αυτά τα ταμεία ασφάλισης, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει και γι' αυτό είμαστε τόσο προσεκτικοί και θα μεριμνήσουμε ώστε να μάθουμε από τις εμπειρίες του παρελθόντος, όπως από αυτά που έγιναν για τους συνεταιρισμούς. Ε, και στις σχέσεις μας με το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά, αν θέλετε, ρηξοί και ε, θα πρέπει να ε, βασιστούμε στην ιστορία. Πάντως η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι πιο ανθεκτικές, είναι πιο βιώσιμες αυτές, πιο βιώσιμα, συγγνώμη, αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης. Και Ε, αυτή η εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν θα μας καθοδηγήσουν στο μέλλον γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και κράτη που δεν έχουν τέτοια ταμεία αλληλασφάλισης. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις παρελθούς εμπειρίες ώστε να βρούμε νέα μέσα και να επιτύχουμε τους απότερους στόχους μας που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική προστασία. Χάρη σε αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης διεκδικώντας εξ ονόματός τους ένα καθεστώς, ευρωπαϊκό καθεστώς. Ως προς το θέμα της ακρόασης, ε, Πρόεδρε, πολύ σημαντικό ε, είναι κατά τη γνώμη μου σε μια ακρόαση να ακούσουμε τους ε, βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που τώρα προωθούμε. και θα μάθουμε από την εμπειρία που είχαν διάφορα κράτη-μέλη στο παρελθόν. Αφήστε που υπάρχουν και συνάδελφοι στους οποίους ε, ακόμη πρέπει να πείσουμε για τα θετικά ε, αυτής της πρότασης, τα θετικά στοιχεία αυτής της πρότασης. Λοιπόν, είναι χρήσιμο το να διοργανώσουμε μια ακρόαση ε, και θα σας υποστηρίξω εφόσον είμαι η συγκήτρια και θα σας υποστηρίξω και για τις αλλαγές ως προς το χρονοδιάγραμμα, όπως λέγαμε νωρίτερα. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει πάρα πολύ άνετο ε, χρονοδιάγραμμα, έχει πάρα πολύ καιρό. Γιατί να μην επωφεληθούμε κι εμείς και να παρατείνουμε από πλευράς μας ε, την ε, ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών πέραν της 10ης Απριλίου. εγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση στην Επιτροπή μας όχι μόνο ενσωματώνοντας αυτή την μελέτη που χρηματοδοτήσαμε και παραγγείλαμε για τα Ταμεία Αλληλασφάλισης αλλά να συμπεριλάβουμε και το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα αναλόγως. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, για να δούμε συγκεκριμένα τι ημερομηνίε. Θα έχουμε το σχέδιο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων τον Ιούνιο, είπαμε. Εξέταση του σχεδίου 9-10 Απριλίου λέει εδώ πέρα στον κατάλογο μου. Άρα, αν τηρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, εμείς θα μπορούσαμε τον Ιούνιο 20 και 21 συγκεκριμένα να διοργανώσουμε αυτή την ακρόαση και την ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες να την ε, θέσουμε σε 11 Ιουλίου, δηλαδή την ε, παύριο μετά την πρώτη εξέταση του σχεδίου στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αλλά μην ανησυχείτε, ούτως ή άλλως θα έχουμε το κείμενο λίγο νωρίτερα στη διάθεσή μας, μετά τροπολογίες 6 ή 18 Σεπτεμβρίου και τα ψηφίσουμε στις 8 ή στις 9 Οκτωβρίου. Πώς σας φαίνεται το νέο χρονοδιάγραμμα. Πολύ ωραία. Θα ενημερώσουμε και τους συντονιστές αλλά δεν διαβλέπω κάποια δυσκολία. Μας, ε, μέσα στα μαύρα σκοτάδια μας έχουν βυθίσει εδώ, αλλά ε, να χαμογελάτε γιατί θα βγούμε και φωτογραφία και πρέπει να φαινόμαστε υπέροχοι. Ξέρετε ότι δεν βγαίνουν καλέ φωτογραφίε όταν έχει πολύ φω, να σηκώνουν και τα στόρια. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και σα δίνω ραντεβού για μια εξαιρετικά σημαντική ανταλλαγή απόψεων κατόπιν αιτήματο τη διάσκεψη των Προέδρων των Ομάδων, που ανέλαβε μια χρήσιμη πρωτοβουλία, διότι στι 5 έχουμε μεικτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για μια ανταλλαγή απόψεων για την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα παρουσία των εκπροσώπων της Τρόικα. Στις 5 ε, η ώρα ραντεβού δύο ρόφους παρακάτω στην αίθουσα 2Q2.